για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 ναι, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συναδέλφισες, ξεκινάμε και πάλι. Θα ήθελα να χαιρετήσω όλους τους συναδέλφους, την Επίτροπο Κρός, να χαιρετήσω και τον εκπρόσωπο